της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λόρδε Χίλ. Ευχαριστώ όλα τα μέλη. Σας ευχαριστώ για την ε, θέλησή σας έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα να απαντήσετε στις γραπτές ερωτήσεις μας και να επανέλθετε ενώπιόν μας για αυτή τη συμπληρωματική ανταλλαγή απόψεων. Τώρα, αν θέλετε παρακαλώ ε, ένα-δυο λεπτά για μερικές ε, καταληκτικές παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, ε, ε, ακούσατε και τον κύριο Κατάινεν ε, πριν από μένα, κάθεστε όλο το πρωί εδώ. Στην τελευταία ερώτηση μου δόθηκε η, ευκαιρία απαντώντας να πω αυτά που ήθελα να πω. Από πλευράς τώρα του χαρακτήρα μου ήθελα να σας πω ότι οπωσδήποτε με ενεργητικότητα, ενθουσιασμό και αφοσίωση και ανεξαρτησία βεβαίω θα ασχοληθώ με τα θέματα αυτά. Και βεβαίως ακαιρεότητα. Το μόνο άλλο που μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες εβδομάδες και ιδιαίτερα το τελευταίο εξαήμερο είναι ότι χρειάζεται αντοχή διότι τις τελευταίες εβδομάδες χρειάστηκε πολύ αντοχή χρειάστηκε να υπερβώ κάποιες, ε, κάποια καχυποψία επειδή είμαι Βρετανός και μάλιστα για αυτήν την ε, αρμοδιότητα. Έκανα ό,τι μπορούσα, ελπίζω να καθησύχασα αυτούς τους φόβους παρά τον ε, περίεργο χαρακτήρα του φλερτ μας μέχρι τώρα ελπίζω να έχω την ευκαιρία από σύντομη σχέση να μετατρέψω τη σχέση μας σε σταθερή και πιο επικερδή και ελπίζω να εργαστούμε μαζί για τα θέματα αυτά την προσεχή πενταετία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος για την αντοχή σας επίσης και για το στυλ σας ε, πέρα στις συνεδριά